Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 86. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 87. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 88 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 127 υπέρ. Συγγνώμη, ψηφίζουμε. Έκλεισε. απορρίπτεται. Η 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 149 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 89 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 90. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 113. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 91. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 130. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 92. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 131. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 132 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Υπάρχει πρόβλημα τεχνολογικής φύσεως. Μπλοκάριζε το σύστημα. Υπομονή παρακαλώ. Δυστυχώς ε, ε, η τεχνολογία μας εγκατέλειψε για λίγο. Λοιπόν, για τεχνικού ε, λόγου ε, πρέπει να ξαναψηφίσουμε για την 131. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 132 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 93. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 94 ψηφίζουμε έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται η 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 ψηφίζουμε έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται 96 ψηφίζουμε Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 97 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 98 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 99 υπέρ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Οι 100 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 101 ψηφίζουμε. Έκλεισε. απορρίπτεται. Η 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 6D υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 11 δι ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε. Απορρίπτεται η 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 13 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται η 14 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται η 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τρίτο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τροπολογία 15. Ψηφίζουμε. Έκλεισε.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 Απορρίπτεται. 29. «29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, η 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, η 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στο πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Και τώρα θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση όσον αφορά το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Κιούσα. Πέρας. Εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 32, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 33. Ψηφίζουμε. Πέρας. Respinto. 118. Απερίφθη 33. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 34. Ψηφίζουμε. Πέρας. Respinto. Απορρίπτεται. Le prima parte chi a favore. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 37. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 37. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 136. Ψηφίζουμε. Πέρας. Respin. Απορρίπτεται. 119. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 38. Ψηφίζουμε. Πέρας.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 αποχές απορρίπτεται 108 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 109 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 45 πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική B. Y. Αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 49 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται όχι απορρίπτεται διορθώνει ο πρόεδρος απορρίπτεται το 49 τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 ψηφίζουμε Πέρασε απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 110. Ψηφίζουμε. Πέρα. Απορρίπτεται. 53. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Με το πέρας των ψηφοφοριών θέλω να σας πω το εξή. Έχουμε κάτι για την έκθεση Αρένα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η θέση της πρώτης ανάγνωσης, η θέση του Κοινοβουλίου. Έχετε κάποια παρατήρηση? Όχι, επομένως. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση και σας ευχαριστώ. Και τώρα, διάλειμμα δύο λεπτών για να περιμένουμε να φύγουν οι συναλληλθοί που θέλουν και κατόπιν θα αρχίσουμε με τις δηλώσεις ψήφου που υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στις δυόμιση ούτως ώστε να τηρήσουμε τις ε, συμφωνίες με τα σύνδικατα. Και τώρα αρχίζουμε με τις ε, ε, αιτιολογήσεις ψήφου. Είπαμε θα πρέπει να δύο δυόμιση ώρα και οι παρεμβάσεις ε, που δεν πρόκειται να γίνουν σήμερα πρόκειται να μετατέθουν για την αυριανή σύνοδο, μετά τις αυριανές ψηφοφορίες. Procediamo con la relazione di Maria και τώρα ξεκινούμε. Έκθεση αρένα όσον αφορά το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Την ε, λόγο έχει ο κύριο Νότιο Μαριά ένα λεπτό. Νότης Μαριά ένα λεπτό. Μαρία, ε, Κύριε Νότη. Κύριε Νότη λέει ο Πρόεδρος. Απλά δεν υπάρχει ησυχία και οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε. Παρακαλώ συνάδελφοι να βγείτε από την, από την αίθουσα για να αρχίσουμε τις αιτιολογήσεις ψήφου. Και έτσι να μην ενοχλούνται οι αγορητές. Ένα λεπτό κύριε Μαριά. Το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει πραγματικά για τη στήριξη της απασχόλησης. Διότι σε μια φάση όπου η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει σε τεράστια ανεργία, σε outsourcing των επιχειρήσεων, σε χτύπημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θεωρώ ότι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης μπορεί να στηρίξει και έχει στηρίξει την προσπάθεια προκειμένου οι άνεργοι να μπορέσουν και να καταρτιστούν και φυσικά να πάρουν μια οικονομική στήριξη. Δυστυχώς στην Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί τα κονδύλια αυτού του ταμείου το οποίο θα μπορούσε να έχει συνεισφέρει πραγματικά για να απαλύνει κάπως την φτωχοποίηση του ελληνικού λαού που έχει επέλθει με τα μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα με τη νέα ρύθμιση θα δοθεί ευκαιρία για περαιτέρω στήριξη και σε σχέση με την ανεργία που δημιουργείται λόγω και των αυτοματισμών και των νέων τεχνολογιών. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο κύριος Χάουαρθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την επιτροπή των Προπολογισμών, πρέπει να σα πω ότι έχουμε εκθέσει και εγκρίνουμε εκθέσει όσον αφορά αυτό το ταμείο όμως κανείς δεν τις λαμβάνει υπόψη αυτές τις εκθέσεις λόγω της ε, ε γιατί έχουμε τόσο κόσμο που απολύεται, έχουμε τόσους υπεράριθμους ε, Είδατε τι γίνεται και στη Γαλλία, στη Νόκια, στη Φιλανδία, τι γίνεται στον κλάδο λιανική, στην Ελλάδα, στα, επίσης στο Γλωσσοφαντουργία, στην Πορτογαλία. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ε, δώσει χέρι αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το νέο MFF δώσει 1,6 δι. Ε, σε μία σειρά ετών. Οπότε κατά αυτόν τον ε, τρόπο δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι θετική αυτή η έκθεση να διευρυνθεί το πεδίο δράσεως του Ταμείου, να αυξηθεί η χρηματοδότηση, γιατί από το 2007 τον Ιούλιο είχαμε 161 περιπτώσεις από 21 κράτη-μέλη. Ε, δυστυχώς όμως η Βρετανική κυβέρνηση δεν συμμετέσχε σε καμία από τι σχετικέ ενέργειες και πρωτοβουλίε. Ευχαριστώ πολύ. Πάλμερ, ένα λεπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, στην ιδέα για αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης θα βοηθήσουμε τη βιομηχανία, θα βοηθήσουμε κάποιες περιφέρειες να κάνουν το μετασχηματισμό, να ανταποκριθούν στα προβλήματα, στις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας που συνέχεια αλλάζει, συνέχεια μετασχηματίζεται με τεχνολογία, ε, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποίηση, να βγούμε από την ε, οικονομία του άνθρακα. Αλλά θα πρέπει να διδαχθούμε από την πρόσφατη ιστορία, συναδελφοί. Είδατε τι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολλά μέρη, όπου χάσαν καλές δουλειές, καλοπληρωμένες, ε, στα ανθρακοριχεία, στα χαριβουργία και αντί αυτών τώρα υπάρχουν κάποιες ευάλωτες δουλειές με αυτές τις συμβάσεις μηδενικών ορών πολύ χαμηλή μισθή. Άρα με τέτοια ταμεία όπως το εν λόγω ταμείο ε, έχουμε κάτι θετικό, οπότε παρακαλώ όλοι, όλοι οι συνάδελφοι να μην δημιουργούμε μόνο θέσει εργασία. Θα πρέπει να προσέχουμε και τι είδου θέσει απασχόληση ε, θεσπίζουμε. Θα πρέπει να είναι θέση εργασία αξιοπρεπή. Ο πρόεδρο. Μα κινείς έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αποτέλεσμα αυτών των αναδιορθώσεων στι εταιρείε έχουμε πάρα πολλού εργαζόμενου σε κίνδυνο αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι αρνητικό η παγκοσμιοποίηση, γιατί προσφέρονται πάρα πολλέ ευκαιρίε που δεν είχαν οι πατεράδε μα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι περισσότερη ελεγγύη. Ευχαριστώ στην Μαρία Ρένα από το Βέλγιο. Γιατί το πνεύμα το σωστό διαπνέει το κείμενο, έχουμε ενέργεια, τεχνολογία, το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι θέματα παγκοσμιοποίηση και έχουμε προστιθέμενη αξία στην πρόταση τη Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, η αντιμετώπιση τη παγκοσμιοποίησης δεν γίνεται χωρί να γίνει προσαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γίνεται στη χώρα μου, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, έχουμε αλλαγέ, αλλάζει η αγορά εργασία, ταχύτατα. Και το Βαλτικό Κέντρο για Ερευνητική Δημοσιογραφία λέει ότι σχεδόν η μισή στη Λετωνία ε, θα είναι πάνω από 50 μέχρι το 2030. Άρα να βοηθήσετε τη χώρα μας ε, όσο γίνεται πρόεδρος. Κλούνε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την έκθεση σχετικά με το Παγκοσμιοποιημένο Ταμείο. Ε, είναι πολύ σημαντικό για όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης ε, και λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Θα ήθελα να χαιρετήσω ιδιαίτερως κάποιες διατάξεις που προτείνονται έτσι ώστε να περιοριστούν περιστεί ο αριθμό των ε, απολυμμένων από 500 σε 200. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μικρέ χώρε όπω είναι η Ιρλανδία, αλλά και για τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, το Ταμείο τη Παγκοσμιοποίηση είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ιρλανδία. Έχει οδηγήσει σε 10 προγράμματα που έχουν εγκριθεί και έχει χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση της σύμβασης με την Lufthansa. Πράγματι συμπληρώνει τα εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως και οι συνάδελφοί μου, ε, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω αυτήν την έκθεση και, να, και εύχομαι η συγήτρια. να επεκτείνει και να ε, παρατείνει αυτήν την ε, ρύθμιση Έχουμε τώρα 145.000 ε, ε, ανέργους, πρέπει να τους δοθούν νέες θέσεις απασχόλησης, νέα εκπαίδευση, να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να ανοίξουν τη δική τους τη δουλειά. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ε, συστήσω τη μείωση από 500 σε 200, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανώτατα στελέχη που χάνουν τη θέση τους να βρεθεί κάποια λύση. Είναι ένα θαυμάσιο ταμείο και πραγματικά δείχνει ότι η καρδιά της Ευρώπης εξακολουθεί να πάλεται. Επόμενη ομιλία, το κύριος, ε, επόμενη ο κύριος Μαριάς. Και η βία, η δημοσιονομική προσαρμογή έχουν γεμίσει την Ευρώπη με στρατιές ανέργων, και εκατομμύρια φτωχούς. αυτή η πολιτική δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και τα όποια μέτρα έρχονται να προσθεθούν για να απαλύνουν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής μέσω του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου δεν μπορούν να χτυπήσουν το κακό στη ρίζα του. σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα κονδύλια του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου plus να αξιοποιηθούν από τις περιφέρειες να αξιοποιηθούν από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου να πάνε πραγματικά για τη στήριξη της κατάρτισης της επιμόρφωσης να στηρίξουν κυρίως τους μακροχρόνια ανέργους να στηρίξουν επίσης τη φτώχεια η οποία χτυπάει την ευρωπαϊκή ένωση να γίνουν πάρα πολλές δράσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους μέτρα οποία και κονδύλια τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα κράτη μέλη. Ιδίω οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου που έχουν χτυπηθεί από τα μνημόνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ διότι υπάρχουν κοινωνικές προκλήσεις. Αντιμετώπιση της ανεργία των νέων, διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων ε, και αγοράς εργασίας, αυτά πρέπει να αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απειλείται από όλες αυτές τις πιέσεις. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις ανισότητες αφού το θέσουμε αυτό ως προτεραιότητα. Τα μέτρα τα οποία προτείνονται θα πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά, γιατί η παιδική ένδυα επηρεάζει πάνω από τα μισά παιδιά στη Βουλγαρία. Δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Πολύ ανησυχητικές ενδείξεις. Και είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ευημερία για τους νέους. Μαμίκινς, Αντρέης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεγάλο πλεονέκτημα της έκθεσης αυτής είναι ότι τα κράτη-μέλη μπορούν με ευέλικτο τρόπο να κατευθύνουν τα χρήματα στα πιο επίγοντα θέματα, αγορά εργασίας, η κοινωνική προστασία, η προστασία της υγείας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κέρια σημασία η Επιτροπή να έχει την εποπτεία του πώ και πού δαπανώνται τα χρήματα αυτά. Και το λέω αυτό διότι ορισμένε χώρε όπω η Λετωνία έχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Στη Λετωνία η ρωσόφωνη μειονότητα είναι 24% του πληθυσμού και δεν τη επιτρέπεται να έχει ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση στη ρωσική γλώσσα. Και μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από το Σεπτέμβριο του 2019 τα παιδιά δεν θα μπορούν να πάνε σχολείο στη μητρική του ε, ρωσική γλώσσα. Όλα αυτά είναι σαφείς ενδείξεις ότι οι νέοι δεν μπορούν ε, να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα, να έχουν σωστή εκπαίδευση λόγω της περιοριστικής γλωσσικής πολιτικής και αυτό πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ. Πάλι με ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Την προηγούμενη φορά που ε, το εξήτασα δεν υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι τα σούπερ μάρκετ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλά εξοπλισμένα. Αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι όλο και μεγαλύτερες ουρές υπάρχουν ε, για συσίτια και για προσφερόμενα γεύματα, πολλά από τα οποία προσφέρονται με χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτή τη φτώχεια και την έλλειψη τροφίμων για τους στοχούς πληθυσμούς είναι όχι να ασχολούμεθα με τους εκατομμυριούχους ε, που δεν θα πληρώσουν το τίμημα του Brexit, αλλά να ασχολούμεθα με αυτούς που θα πληγούν από την έλλειψη συμφωνίας για την ε, οργανωμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει καν η πιθανότητα μη συμφωνίας για τον Brexit. Ευχαριστώ. έτσι ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν συμφωνώ με την πρόταση του να συρρυκνωθούν οι επενδύσεις για το Ταμείο επενδύσουν για αυτά τα 7 δις ευρώ η πρόταση του Κοινοβουλίου πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μιλάει για αύξηση κατά 106 δις ευρώ. Πρόκειται για ένα μέσο σημαντικό για κατάρτιση, εκπαίδευση, για νέες μορφές απασχόλησης, ιδίως για τους νέους. Και επίσης είναι και ένα μέσο βελτίωση της ζωής αυτών που έχουν αναπηρία, όλων των περιθωριοποιημένων όλοι τώρα μπορούν να ενταχθούν πιο πολύ στην κοινωνία. Κατά πολέμηση επίσης της φτώχειας. Έτσι, επίσης χτυπάμε και την φτώχεια των ανηλίκων. Άρα περισσότεροι πόροι χρειάζονται, περισσότερες δραστηριότητες για τις νέες μορφές γνώσης. Ευχαριστούμε κυρία Κλούνε τώρα ένα λεπτό. Θετική σημερινή πρόταση να ενισχυθεί το Ταμείο για την επόμενη περίοδο μέχρι το 27. Τώρα το Κοινωνικό Ταμείο θα επιστρατεύσει αυτή την ε, πρωτοβουλία νέους πόρους ε, για τους ε, μη προνομιούχους και έτσι θα έχουμε αυτή την κοινωνική πρωτοβουλία για την ανεργία, θα έχουμε περισσότερη απασχολησιμότητα και θα πλήξουμε την φτώχεια αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό θα προσέξουμε ιδίω ε, τους νέους και τους ανηλίκους. Επομένως, πρόκειται για ένα ταμείο που αξίζει. Ε, αφορά ε, τα άτομα, τους ανθρώπους. Ήδη είπαμε ότι στα πλαίσια πραγματοποίησης θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, τα προβλήματα και πρόκειται επίσης για βοήθεια προς την ισόβια κατάρτιση. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε να συνεχίσουμε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συν να το υποστηρίζουμε και να υπάρχει θετική επίπτωση άμεσα στις κοινότητες Σουίτσα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι θετική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2021 21 έω 27 πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν αφορά μόνο την απασχόληση και την ε, κοινωνική ένταξη. Το κοινωνικό ταμείο συνεχίζει να δράει για την πολιτική συνοχή. Συνεχίζει να βοηθά την πρωτοβουλία για τους νέους και άλλα προγράμματα σε σχέση με την Επιτροπή, με την στρατηγική συνοχή. Τώρα έχουμε 106 δις ευρώ που θα πρικοδοτήσουν που είναι αρκετό όσον αφορά το 27% της πολιτικής της συνοχής. Άρα είναι θετικό. Και να έχουμε και κάποιο είδους απλούστευση στη διαδικασία κατανομής των ε, πόρων και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα θετικό βήμα. Άρα είμαστε υπέρ του Ταμείου αυτή. Νικόλα το ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για το Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ για την περίοδο 21-27 να συνεχίσει να βοηθά στην απασχόληση, στην κοινωνική ένταξη και ε, να γίνουν βήματα προς τα εμπρός ώστε να υλοποιηθεί η κοινωνική διάσταση, να συνεχίσουν να έχουμε στόχο την κάλυψη των ε, νέων. Υπάρχει πρόβλημα ε, ανεργίας για τους νέους, οπότε αυτό το ταμείο θα πρέπει να έχει ε, μέτρα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των ε, νέων, να προσέξουμε ιδίω αυτούς που δεν είναι δραστήριοι, είναι μακριά από την αγορά απασχόλησης. Το ταμείο αυτό να χρησιμοποιηθεί για την αγορά απασχόλησης, να εξυγχρονίσει την, ε, στις δημόσιες ε, υπηρεσίες απασχόλησης και επίσης και τον ε, επαγγελματικό προσανατολισμό να δούμε τι θα γίνει για τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό ανησυχεί. Άρα χρειάζεται αυτό το ταμείο να δώσει μεγάλη πρικοδότηση για καταπολέμηση της φτώχειας και υπέρ της κοινωνικής ένταξης. Ευχαριστούμε κύριε Καπούτο. Και τώρα Πασκάλ Άρημο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρά λοιπόν ε, την ιδιαίτερα απογοητευτική στάση στην ψηφοφορία στις, ε, στα δύο θέματα που ε, κατατέθηκαν, Εμεί θέλουμε να πούμε ότι το κείμενο τη Ρέτζι είναι ικανοποιητικό και γι' αυτό υπερψηφίσαμε. Γιατί καταβάλλονται προσπάθειε ε, να υπάρχει μια μεικτή αρχιτεκτονική δομή. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον νέο κανισμό περιλαμβάνει βέβαια διάφορα κρίσιμα θέματα. Εμεί ε, παρεμβήκαμε σε όλε τι φάσει και έτσι λοιπόν πρόκυψε ένα κείμενο πολύ ικανοποιητικό όπως ψηφίστηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα ε, διασυνοριακά προγράμματα, η αλλαγή της αρχιτεκτονικής δομής ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θαλάσσια συνεργασία. Αυτό δεν μπορούσε να στηριχθεί όχι μόνο στις περιφέρειες αλλά και γενικότερα για να υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή. Θα έπρεπε να υπάρχουν ουσιαστικέ αλλαγέ ε, ουσιαστικές αλλαγές στα, θαλάσσια, στα θέματα θαλάσσια συνεργασία. Προβλέπονται 11 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το συνολικό ποσό, και περίπου ένα δις ε, για κάθε νέο εργαλείο για να υπάρξουν καινοτομίες. Έχει αυξηθεί το επίπεδο συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80% έχουν υπολογιστεί διαφορετικά οι συνεισφορές. Έτσι λοιπόν εναπόκειται στις ε, τοπικές αρχές να έχουν την απαραίτητη ρευστότητα για να ξεκινήσουν προγράμματα στην επικράτειά τους. Θα θέλαμε να επενθυμίσουμε ότι όλα τα στοιχεία του Ιντερεκ θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους της ε, χιλιετίας, δηλαδή ε, θα πρέπει να ενισχυθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις ως εκ τούτου θεωρούμε ότι ο πέμπτο πυλώνα θα πρέπει να εστιάζει στο να υπάρχουν σχέσει ανάμεσα στις περιοχές που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες με εκείνες που είναι ανεπτυγμένε. Ε, οικοσυστήματα καινοτόμα, λειτουργικά, έτσι ώστε να καλυφθεί το gap, το κενό ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες και μέσα στα κράτη και διεθνικά. Σα ευχαριστώ πολύ. Περιφερειακής ανάπτυξης, όπως ξέρουμε, στηρίζει τις περιφέρειες και βεβαίως το πρόγραμμα interreg απεδείχθη πολύ σημαντικό για την ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων κρατών μελών τα οποία γυτνιάζουν. ταυτόχρονα όμως η γυτνίαση ορισμένες φορές μπορεί να αποβεί και αρνητική για ορισμένες οικονομίες διότι έχουμε κράτη όπως είναι η βουλγαρία στην οποία υπάρχει χαμηλή φορολογία και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για τον ομό εύρου δράμας και σερών που γυτνιάζουν με τη βουλγαρία και έτσι δημιουργείται θα έλεγε κανείς ένα φορολογικό ντάμπινγκ γι' αυτό πλέον το interreg πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να στηρίξει εκείνες τις οικονομίες οι οποίες υφίστανται ένα αθέμητο ανταγωνισμό από γειτονιάζουσες χώρες και να βοηθηθούν πλέον οι χώρες όπως είναι η ελλάδα προκειμένου να στηριχτούν οι οικονομίες να στηριχτούν οι επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται ένα αθέμητο ανταγωνισμό λόγω της γειτονίασης με τη βουλγαρία η οποία πραγματικά κάνει ένα φορολογικό dumping με πολύ φτηνό και χαμηλό ΦΠΑ αλλά και φορολογία εισοδήματος. Ευχαριστώ. Τα προγράμματα Interreg είναι πολύ σημαντικά διότι ενισχύουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ιδίω η πρώτη συνιστόσα της διαμεθοριακής συνεργασίας. Χαίρομαι λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε την αύξηση χρηματοδότησης για την διασυνοριακή συνεργασία. Τα κονδύλια για τη διασυνοριακή χρηματοδότηση είναι τώρα υψηλότερα από ό,τι στην αρχική πρόταση τη Επιτρο... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 11 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύονται σε τέτοια προγράμματα. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δαπανώνται αποτελεσματικά και με όσο δυνατόν πιο απλουστευμένες διαδικασίε. Χαίρομαι λοιπόν διότι πολλέ τροπολογίε που κατέθεσα για την απλούστευση τη διαδικασία έχουν γίνει αποδεκτέ. και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε μικρότερο διοικητικό φόρτο για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είχαν υποδείξει οι δικαιούχοι. Και το, θέμα, το πρόγραμμα της καινοτομία είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι κατά 0,3% θα αυξηθεί το κονδύλι για την καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ, Σβίτσα. Ενδιαφέρομαι για το θέμα αυτό από τότε που ήμουν σκιώδης εισηγήτρια για την Επιτροπή ΑΦΕΤ για το αντίστοιχο θέμα. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης που ασχολήθηκαν με το φάκελο αυτό και που βοήθησαν να αναδείξουμε τη σημασία αυτού του θέματος. Θέλουμε να μειώσουμε την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, να γίνει πιο εύκολη η χρηματοδότηση και χαιρόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για το Interreg για τη χρηματοδότηση διασυνοριακής συνεργασίας. Συνήθως πρόκειται για μικρά έργα μεταξύ πολιτών και λοιπόν την έκθεση αυτή και ελπίζω ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη χρήση των κονδυλίων, μείωση των διοικητικών φραγμών και όλα αυτά τα έργα θα είναι προ όφελο των πολιτών μα. 11 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι μικρό ποσό. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για το έργο που έχει επιτελέσει. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε την έκθεση για τα φυτοφάρμακα. Πρώτος είναι ο κύριος Νέκοβ για ένα λεπτό. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Είναι σαφές το μήνυμα σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την έγκριση των φυτοφαρμάκων. Τα πράγματα δεν μπορεί να συνεχίσουν να είναι όπως είναι σήμερα. Να υπάρχει 100% διαφάνεια στην έγκριση. Για να μην έχουμε ένα νέο Dwayne Johnson. Να μην έχουμε καρκίνους θα πρέπει να έχουμε νέες μεθόδους προστασίας των φυτών. Πολλά από τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και για την βιοπικιλότητα. Κινδυνεύουν πολύ οι μέλισσες. Άρα με σοβαρότητα να καταπολεμήσουμε τις ε, παράνομες εισαγωγές φυτοφαρμάκων. Πιο αυστηρή έλεγχη στα βουλγαρικά σύνορα. Αυτό θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ θετικό θεωρώ το ότι έχουμε συμμετάσχει ε, στις σχετικές ε, εργασίες για την Ειδική Επιτροπή και έτσι ναι, ως ε, Γκουε έχουμε συμβάλει σε αυτήν την έκθεση και είμαι ικανοποιημένη για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφορία. είναι βήμα προς τα εμπρός. Πάμε για περισσότερη διαφάνεια γιατί τα πράγματα όπως λέει και η Εύσα για τη γλυφοσάτη είναι ανησυχητικά. Οπότε τώρα κάνουμε ό,τι κάναμε και στην εκστρατεία Stop Glyphosate βήμα προς τα έμπρος και ότι η γλυφοσάτη είναι επικίνδυνη χημική ουσία, ε, χτυπάει τα φύτα ε, και άλλους οργανισμούς. Ούτε διαλύεται εύκολα και στην Απουλία, την πατρίδα μου, έχουμε πάρα πολύ γλυφοσάτη στο έδαφος και υπάρχει και ο νόμος Μαρτίνα για τα φυτοφάρμακα και επιτρέπει την έγκριση τέτοιων φυτοφαρμάκων. Άρα τώρα με την σχετική διαδικασία κάνουμε μόνο προς τα εμπρός. Ένα λεπτό η Εύη. Και εγώ, Πρόεδρε, θεωρώ θετικό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της έκθεσης. Είναι σημαντική έκθεση για την έγκριση φυτοφαρμάκων. Έτσι η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε αυτό που θέλουν τόσα εκατομμύρια Ευρωπαίων. Θέλουν αυτά τα τοξικά επικίνδυνα προϊόντα για περιβάλλον, για υγεία, για βιοπικιλότητα, όλα αυτά τα χημικά να απαγορευτούν. Έχουμε τώρα όλες αυτές τις ε, μελέτες, τις ε, δημόσιες, τις διαφανείς διαδικασίες και έτσι θα έχουμε κάποια εγγύηση ότι δεν θα έχουμε άλλη Monsanto Papers, δεν θα έχουμε άλλο σκάνδαλο όπως με τη γλυφοσάτη. Θα προσέξει η Ευρώπη μόνος έτσι περιβάλλον και υγεία. Γκούντα. Ένα λεπτό. Η έκθεση αυτή για την, έκθεση, για την έγκριση των φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άμεση σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Έγκρισης ε, ε, τη ασφάλεια Ασφάλειας των Τροφίμων. Τα έγγραφα σχετικά με τη Μονσάντο έχουν δείξει ότι μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις και σφάλματα σε όλο το σύστημα. Μετά από εννέα μήνε λειτουργία τη Ειδική Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλήγουμε σε ένα μέτριο κείμενο. Ανταποκρίνεται οριακά στι προκλήσει ε, για ε, την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιε πρόοδοι, οι οποίε θα είναι καθοριστικέ ε, για να δημιουργήσουμε στη συνέχεια διαδικασίε έγκριση φυτοφαρμάκων που θα είναι ενδελεχέστερες θα πρέπει να υποχρεώσουμε την Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων ε, να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μορέλ, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψηφίσαμε συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων ανείχνευσης και απαγόρευσης επικίνδυνων φυτοφαρμάκων. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνούμε ότι είναι θετικό βήμα. Παράλληλα όμως, ταυτόχρονα, τα μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι ένα από τα Ινστιτούτα που εργάζονταν για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων είχε αντιγράψει ένα μεγάλο τμήμα των εκθέσεων της Μονσάντο, που είναι ο κατασκευαστής γλυφοσάτης για την οποία όλοι έχουμε τονίσει πόσο επικίνδυνη είναι. Μιλάμε λοιπόν για ένα σκάνδαλο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Θα πρέπει να, ε, να δείξουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και θα πρέπει ε, να πούμε και προς τον αρμόδιο επίτροπο και προς τον υπεύθυνο της ΕΦΣΑ ε, ποια είναι η πραγματικότητα για να μπορέσουμε να έχουμε αξιοπιστία. Καταλαβαίνουμε τα σχετικά με την απαγόρευση κάποιων ε, επικίνδυνων ουσιών, αλλά θα πρέπει και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Κύριος Πόσπισιλ, παρακαλώ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ υποστήριξα αυτή την έκθεση γιατί προβλέπει την ενίσχυση των κανόνων για την ε, αδειοδότηση ε, ζυζανιοκτώνων στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια ποιοτική νομοθεσία για τα 28 κράτη-μέλη. Εγώ υποστήριξα όλες αυτές τις ε, τροπολογίες που προβλέπουν πιο αυστηρή νομοθεσία. Βέβαια, μια τροπολογία που δεν πέρασε είχε ως ε, στόχο να περιορίσει την χρήση των ζανιοκτώνων ε, ε, σε σχέση με τα ζώα. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτή η νέα τεχνολογία θα είναι καλύτερη και χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασε η πρόταση. Χαίρομαι που θα είναι πιο αυστηρές οι προδιαγραφές για την αδειοδότηση νέων ζυζανιοκτών γιατί θεωρώ ότι από αυτή τη νέα καλύτερη νομοθεσία θα υποφεληθούμε όλοι μας. Επόμενη μιλητρία, η κυρία Σουίτσα, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τη γλυφοσάτη. Αυτό οδήγησε στο να υπάρξει επιτροπή ΠΕΣΤΑ, η οποία δούλεψε πολύ σκληρά και αυτή είναι μία από τις ε, εκθέσεις ε, η οποία υποβάλλεται από την αριστερή πλευρά του Κοινοβουλίου και δεν νομίζω ότι ακολουθεί ε, τη σωστή κατεύθυνση έκθεση. Είναι πολύ καλό ότι η φάση διαδικασίας ε, αδειοδότηση έχει δύο φάσεις, η μία σε ενωσιακό επίπεδο και η άλλη σε εθνικό επίπεδο. Ε, έτσι θα γίνεται η αδειοδότηση των προϊόντων προστασίας των φυτών. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση γιατί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο η υγεία των πολιτών μας όσο και το ε, μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος ε, Πόλτσακ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να επιδεικνύει κανείς υπευθυνότητα αλλά και σταθερότητα σε αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάρη όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες, ε, κυρίως στην Τσεχία, η γλυφοσάτη και άλλες ουσίες υπερ καταναλώνονται στη γεωργία και αυτές οι ουσίες κατ' ουσίαν μπορούν να καταστρέψουν οτιδήποτε πράσινο υπάρχει. Ε, θέλω να πω ότι σήμερα στην αγορά υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικέ λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν η αποφάσεις μας θα πρέπει να είναι όσο πιο διαφανής γίνεται. Ε, και πρέπει να ομολογήσω ότι όταν ήμουν στην Επιτροπή Γεωργίας παραπλανήθηκα από μία μελέτη που δεν ήταν διαφανής και θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτή η μελέτη σκόπιμα ε, παραποιήθηκε. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, να υπάρχει διαφάνεια, γι' αυτό είμαι υπέρ αυτής της έκθεσης και ελπίζω ότι η περιβαλλοντική προσέγγιση θα υπερισχύσει στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ και όλους τους ε, συναντέλφου. Λύεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3.